Για μας η συναπόφαση δεν είναι ότι το Συμβούλιο αποφασίζει και το Κοινοβούλιο προσαρμόζεται. Ευχαριστούμε κυρία Γκουλουάρα. Έληξε εδώ αυτή η συζήτηση, θα γίνει αύριο η ψηφοφορία στις 12 και ερχόμαστε τώρα στην επόμενη συζήτηση. Την έκθεση του κυρίου Παλώνε για τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 11 και 12. Θα αρχίσει λοιπόν ο εισηγητής για τέσσερα ολόκληρα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γραμματεία και όλους τους σκιώδεις εισηγητής γιατί είχαμε ουσιαστικά μια αντιπαράθεση μεταξύ καλών ανθρώπων που είχαν κατά νου την κοινή έννοια και δεν ε, είχαν ιδεολογικές ε, προκαταλήψεις. Ε, αν και εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ανησυχητική η κατάσταση. Οι οικονομίες μας δεν βγήκαν ακόμη από την κρίση και το σπιράδι της ύφεσης συνεχίζεται. Έχει καταστροφικό αντίκτυπο οικονομικό η κρίση και έχει δημιουργήσει ανισορροπίες στα δημοσιονομικά και δημιουργεί τεράστιες αποκλήσεις με καταξύ των κρατών μελών και προβλέπεται και κρίση του ΑΕΠ ε, φέτος οι προοπτικές ε, φαίνονται επισφαλείς. Η κρίση έχει μετατραπεί και σε κοινωνική κρίση, αρκεί να δούμε τα στοιχεία σε σχέση με την ανεργία. Εμείς φτάσαμε στο 11% η κατάσταση απαιτεί να ληφθούν επίγοντα μέτρα και η Ευρώπη πρέπει να ξαναρχίσει να αναπτύσσεται. Τα βήματα προ τα μπρο που έγιναν στα πλαίσια τη νέα οικονομική διακυβέρνηση. είναι αξιοσημείωτα. Το Six Pack ευνόησε μια μεγαλύτερη προσπάθεια για την δημοσιονομική εξυγίανση. Έχουμε μια πιο σταθερή χρηματοοικονομική κατάσταση, αλλά αυτό ακόμη δεν αρκεί. Πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων η περίπτωση του ΤΟΥΠΑΚ ε, το υποθύμησε προηγουμένω ε, και ο Επίτροπο. Ε, διέπεται από άλλε διαδικασίε και πρέπει να έχουμε και μία τραπεζική ένωση προκειμένου να έχουμε μεγαλύτερη χρηματοοικονομική δραστηριότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να διερευνήσουμε και άλλου τρόπου διαχείριση τη οικονομική κρίση προκειμένου να ελχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Αλλά αναφεσβήτητα μία μεγαλύτερη αηφορία των δημοσίων οικονομικών είναι το πρώτο βήμα για να συνεχίσει για να αρχίσουμε να αναπτυσσόμαστε η εξυγίανση των δημοσιονομικών είναι η απαραίτητη προπόθεση ε, για την ε, ευρωπαϊκή βελτίωση της οικονομίας και θα πρέπει να υπάρχει αντίκτυπο στους πολίτες και στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Γι' αυτό υπογραμμίζουμε τη σημασία μιας εξυγίανσης που θα βασίζεται περισσότερο στη μείωση των δαπανών και όχι μόνο στη φορολόγηση. Τέτοια μείωση αναφέρεται σε όλα τα κεφαλαία ε, των μη παραγωγικών δαπανών ε, όπως παραδείγματος χάρη και στις ε, δαπάνες, στις μη αποτελεσματικές σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Επίσης είναι σημαντικό να διατηρήσουμε όλα τα παραγωγικά, όλες τις παραγωγικές δαπάνες έρευνα, ανάπτυξη και κατάρτιση και πρέπει να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά κάτι τη φοροδιαφυγή. Εξυγίανση λοιπόν πρέπει να γίνει μέσω της περικοπής των δημοσίων δαπανών, των μη παραγωγικών, ε, παρά επί της αύξησης των φόρων. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε μόνο στο περιθώριο και στην περίπτωση που δεν είναι αρκετέ οι περικοπές των δαπανών. Μέχρι τώρα η αύξηση της φορολογίας ήταν πιο εύκολη για κάποιε κυβερνήσει για να μειωθεί το χρέο στο συντομότερο δυνατό χρόνο όμως αυτό επιτάχυνε την ύφεση. Επομένως πρέπει να ληφθούν σήμερα μέτρα για να μειωθεί ο αρνητικό αντίκτυπος. Μόνο εξυγίανση δεν αρκεί. Μαζί με την εξυγίανση των δημοσίων λογαριασμών οι διάφορες εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ξεκινήσουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις για να ευνοήσουν την οικονομική ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν ε, στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρέπει να βελτιωθεί η αγορά εργασίας μειώνοντας τη φορολογία και θα πρέπει να διευκολυνθούν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και να ε, επιτευχθεί ε, ο ανταγωνισμός που χάθηκε τα τελευταία χρόνια η υπερβολική λιτότητα είχε αντίκτυπο στην κατανάλωση και στις οικογένειες και μείωσε την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και μείωσε τη δραστηριότητα της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστούμε τον κύριο Σεγητή, κύριο Επίτροπος. Εσείς έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Παλώνε και την Επιτροπή, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για αυτή τη σημαντική έκθεση. Καταλαβαίνω ότι η συζήτηση ήταν πολύ έντονη. Αυτό γιατί είναι βαθιά και η κρίση που πλήττει την Ευρώπη και που αναλύει αναλύουν οι εκθέσεις και ανακοινώσεις της Κομισιόν από το 11 και το 12. Σημειώνω δε όντως ότι το σχέδιο ψηφίσματος καταλήγει ότι για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των δημοσίων επενδύσεων και των δημοσιονομικών ότι αυτό είναι απόλυτο στόχος και το περιγράφει και όλες τις προσπάθειες που έκανε η Ένωση τα τελευταία χρόνια για να βελτιώσει την διακυβέρνηση της οικονομική και χρηματοπιστωτική. Ξέραμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να συνεχιστούν και με τρόπο που να χωρίζεται αναχώρα με στόχο να διατηρηθεί η ανάπτυξη και η ισότητα και η ισοπολιτεία μεταξύ των πολιτών. Αυτό συμφωνεί και με την άποψη της Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή μας για την ανάπτυξη του περασμένου Νοεμβρίου. Εάν λοιπόν εγκριθεί η έκθεση αυτή θα ήθελα να σας πω ότι μερικά από τα αιτήματά της έχουν ήδη πληρωθεί στην πράξη, εφαρμοστεί. Ιδιαίτερα η Κομισιόν έχει ήδη συγγράψει ανάλυση ανά χώρα και κάνει σχετικές συστάσεις στην καθεμία. Αναλύει την Ευρωζώνη γενικότερα και δημοσιεύει τις αξιολογήσεις της τακτικά. <coughs> Κυρίες και κύριοι, τους επόμενους μήνες, οι επόμενοι μήνες θα είναι ακόμη δύσκολοι, διότι η οικονομία παραμένει αδύναμη και οι πολίτες ακόμη αισθάνονται το αντικριπό τον αντίκτυπο της κρίσης. Αλλά υπάρχουν και σημεία δείκτες σταθεροποίησης και μεγαλύτερης και αύξησης της εμπιστοσύνης στις αγορές. Πράγμα που φαίνεται από την μείωση των επιτοκίων στην Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία. Η εμπιστοσύνη έχει προωθηθεί και σε ενωσιακό επίπεδο και σε πολλές χώρες μεμονωμένα. Και αυτό φαίνεται από εκθέσεις των κεντρικών τους τραπεζών. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα ελλείμματα έχουν μειωθεί από πάνω το 6% το 9 ή 10 στο περίπου 3% πέρυσι και θα μειωθούν μάλλον κι άλλο προς το 2% φέτος. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όλων όσων έχουν γίνει για την ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης από κοινού από την Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Δεν υπάρχουν λοιπόν τόσο πολλοί λόγια πεσιοδοξίας τώρα όσο πέρυσι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μειώσουμε την προσοχή μας γιατί πρέπει να συνεχίσουμε την εξισορρόπηση των προσπαθειών μας με τους στόχους μας. Και γι' αυτό ακριβώς προτείνουμε αυτό το blueprint για μια βαθύτερη και αληθινότερη οικονομική ένωση και νομισματική που να μπορεί να δώσει σταθερότητα και απασχόληση στους πολίτες που είναι και ο στόχος μας ο επίσημος για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και γι' αυτό καταλήγω ότι για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον δρόμο αυτόν επαναλαμβάνω ότι συμμερίζομαι την έκκλησή σας για την έγκριση προτάσεων όπως την Δήμετρο γιατί η έγκρισή του εξαρτάται από τις αποφάσεις όλων των παραγόντων μεταξύ των οποίων φυσικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις ε, πολιτικές του ομάδες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Τώρα οι ομάδες. Ο κύριος Καράσια από το ΕΛΚ πρώτος. Ναι. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω κάτι εκτός της ημερήσιας διάταξης. Εάν παίρνουμε σοβαρά αυτά τα μέτρα, κύριε Επίτροπε για τα νομισματικά, τότε είστε εσείς ο σωστός υποψήφιος για την Προεδρία της Ευρωζώνης και για πρώτος Υπουργός Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε πρέπει να ενισχύσουμε την Κομισιόν και τον Επίτροπο στον έλεγχο των δημοσίων οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα δεν είναι μόνο να δούμε την σχέση των δημοσιονομικών πολιτικών ε, των κρατών μελών με την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό ένα νέο πρίσμο, αλλά απαιτείται επίσης επιγόντως να αλλάξει η σχέση των προπολογισμών με τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Ναι, επιτύχαμε πολλά, αλλά όχι αρκετά. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία συμφωνήσαμε ευρωπαϊκά εξάμεινο, six-pack, two-pack, δημοσιονομικό σύμφωνο. Όλα αυτά είναι κομμάτι της του απαραίτητου και ενισχυμένου συντονισμού των ε, δημοσιονομικών πολιτικών. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ορμή που αποκτήσαμε για να περάσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές βελτιώσεις ε, για να συμμαζέψουμε τους προϋπολογισμούς. Δεν είναι λογικό να, όπως είπα να, να κοιτά μόνο τα οικονομικά του κεντρικού κράτους και να μην ασχολούμαστε καθόλου με το τι γίνεται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Χρειάζεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έλεγχος των ταμείων με ε, όπως είπα πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί άμεσα. Είναι καλή η έκθεση αλλά πρέπει να δοθεί συνέχεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ποδηματά για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θεωρώ ευτυχή σύμπτωση το γεγονός ότι συζητάμε την έκθεση του κυρίου Παλώνε για τα δημόσια οικονομικά σήμερα την ίδια μέρα δηλαδή με την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με την συμμετοχή του αυστριακού καγκελάριου του κυρίου φάιμαν για το μέλλον της ευρώπης γιατί αυτό που αναδείχθηκε από την πρωινή συζήτηση είναι ότι εάν θέλουμε να έχει μέλλον η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να ξαναφέρουμε τους πολίτε στο προσκήνιο με περισσότερη και με καλύτερης ποιότητας δημοκρατία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη με καταπολέμηση όλων των ανισοτήτων με προστασία της κοινωνικής συνοχής και με περιφρούρηση του κοινοτικού κεκτημένου σε όλα ανεξαιρέτως τα επίπεδα και στο κοινωνικό και στο περιβαλλοντικό και όχι μόνο στο δημοσιονομικό. και αυτό σημαίνει στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια δημοσιονομικά προγράμματα φιλικά προς την ανάπτυξη και προγράμματα διαρθρωτικών αλλαγών που σέβονται και δεν αποδομούν τα κοινωνικά δικαιώματα που προάγουν τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα και διαφυλάττουν το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. κύριε επίτροπε γνωρίζοντας ότι γνωρίζετε πως ορισμένες χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής δεν βρίσκονται σε αυτή την ισορροπία που περιέγραψα σας ζητώ να κινητοποιηθείτε και να παρέμβετε για να προσπαθήσετε να την εξασφαλίσετε γιατί αυτό είναι ο μοναδικός δρόμος και για να έχει μέλλον η ευρώπη και για να μην καταλήγουμε διαρκώς στο ίδιο σημείο αμφισβήτησης της βιωσιμότητας των δημοσιονομικών και μακροοικονομικών προοπτικών της ευρωζώνης αλλά και συρρήκνωσης της εμπιστοσύνης των πολιτών. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ποδηματά. η Μπαρσέλης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πίτροπε. Πώς να φροντίσει κανείς τη δημοσία οικονομικά για να είναι βιώσιμα είναι το κύριο πολιτικό και οικονομικό ζήτημα αυτής της δεκαετίας. Για να πετύχουμε τον στόχο αυτό, οι ομάδες του, αυτού του κοινοβουλίου πιστεύουν ε, ότι είναι πιο αποτελεσματική η περικοπή των δεκανών ε, παρά φορολόγηση. Αν ε, κατευθυνόνται προς την ανάπτυξη αυτή η έκθεση τονίζει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον υπάρχουν δύο πολύ ενδιαφέρουσες ιδέες που θα ήθελα να επισημάνω. Καταρχήν, αυτό το κοινοβούλιο δηλώνει ότι οι περιφερειές χωρίς καμία ευθύνη για τα έσοδα που χρησιμοποιούνται μόνο από μεταβιβάσεις της κεντρικής κυβέρνησης ε, είναι πιο πιθανό να αποτύχουν στις προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης αυτή η χρηματοδότηση για τις περιφέρειες ε, πολύ μακριά από το φορολογικό φεντεραλισμό είναι κακή για όλους ε, τελικά ε, κάνει τις περιφέρειες να δεν τους ίδιους, τους ίδιους πόρους της και συμβαίνει αυτό σήμερα στην Ισπανία. Δεύτερη ιδέα τα Υπουργεία ε, και τα τμήματα της κυβέρνησης που δεν έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες θα πρέπει να καταργηθούν. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε προσπάθειες ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης ενώ διατηρείται μια άχρηστη γραφειοκρατία. Στην Ισπανία, παραδείγματο χάρη, γιατί χρειαζόμαστε το Υπουργείο Υγεία και το Υπουργείο Παιδεία και το Υπουργείο Πολιτισμού όταν όλε οι αρμοδιότητε του τομεί αυτού ε, είναι στο επίπεδο των περιφερειών λοιπόν και αγαπητοί συναδελφοί, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παλαιόνο για την πολύ καλή δουλειά του. Την πολύ καλή δουλειά του. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Έχουτ από την ομάδα των Πρασίνων. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο Παλόνι για την καλή συνεργασία για την έκθεση αυτή για τα δημόσια οικονομικά και όλους τους κοιόδης εισηγητές που δίνει νομίζω μια ισορροπημένη εικόνα για το που βρισκόμαστε. Και νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά τα δημόσια οικονομικά, να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις και να σταματήσουν οι επενδύσεις σε μη παραγωγικούς τομείς. Σωστό αυτό, αλλά αναφέρεται πως έχουμε προβλήματα στην Ευρωζώνη. Δεν θα αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου η οικονομία το 2013 και αυτό οφείλεται και στην ατζέντα των προηγουμένων ετών με την πολύ αυστηρή λιτότητα. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην ε, εξοικονόμηση αλλά και στις επενδύσεις για το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία στην Ευρώπη για να υπάρξει μια διαρκής και αηφόρος ανάπτυξη. Και άρα απευθύνομαι εδώ πέρα στον κύριο Ολιρέν, ο οποίος λέει πως αυτά τα ενσωματώνουμε και βεβαίως είναι η συνέχεια των όσων κάνει η Κομισιόν. Εγώ διαβάζω άλλα πράγματα στις συστάσεις της Κομισιόν και ε, στην έκθεση αυτή ζητάει εδώ πέρα ξεκάθαρα το Κοινοβούλιο μετατόπιση των φόρων από την εργασία στο περιβαλλοντικό κόστος. Πού φαίνεται αυτό Πού το βλέπουμε αυτό στις στάσεις Κομισιόν. Πού βλέπουμε η Κομισιόν να λέει κάτι για τη φοροδιαφυγή. Πού λέμε κάτι, πού κάνετε κάποια σύσταση για τις επενδύσεις. Μπορούν να γίνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα και η έκθεση αυτή σας δείχνει πως η Κομισιόν δεν έχει κάνει όλα όσα πρέπει. Ναι, μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αλλά τώρα πρέπει να ασχοληθείτε με τη φοροδιαφυγή, μετατόπιση των φόρων από την εργασία στο περιβαλλοντικό κόστος, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να πείτε. Αυτά θα ήθελα να ακούσω από τον Επίτροπο. Ο Στρέτζεκ ε, από το ECR για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε αυτή την ολομέλεια ε, συνήθως ασκώ κριτική, αλλά για μία φορά έχω την ικανοποίηση να πω ότι η έκθεση του κυρίου Παλών ε, περιλαμβάνει μία σειρά θετικών ωφέλιμων στοιχείων και περιλαμβάνει μία σειρά πυλώνων που υποστηρίζουμε και μάλιστα θα πρέπει να χαιρετήσουμε και πολλά από αυτά τα στοιχεία. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ, το χάρη, το ότι αναφέρεται το ότι πρέπει οι κρατικές μεταρρυθμίσεις ε, να έχουν ε, στόχο να καταργήσουν όλα ε, τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Εγώ νομίζω ότι πολλές φορές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριφέρεται με πολύ γραφειοκρατικό τρόπο. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτό που λέτε. Επίσης, ο κύριος Παλώνε αναφέρεται στο να ε, καταργηθούν ε, κάποιοι φορείς που δεν έχουν αρμοδιότητα σε κρατικό επίπεδο και αυτό σημαίνει ότι χάνονται πάρα πολλά χρήματα. Αυτή η απέτηση να ε, Έχουμε επίση βελτίωση των προσόντων ανάλογα με τι ανάγκε τη αγορά εργασία. Είναι επίση κάτι πολύ θετικό όμω. Εγώ νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι και η παρατήρηση του κυρίου Παλώνε όπου αναφέρεται στην εργασία που δεν αμείβεται όπως πρέπει και ε, πιστεύω ότι πολύ θετικό είναι και το στοιχείο που αναφέρεται στα φορολογικά έσοδα. Όλα όσα θα θέλαμε εμείς συντερτικοί υπάρχουν στην έκθεση αυτή. Μεγαλύτερος ανταγωνισμός, ε, μικρότερη ρύθμιση, μεγαλύτερος ρόλος του ιδιωτικού τομέα. Εγώ νομίζω ότι στο μέλλον μπορούμε να εμβαθύνουμε ακολουθώντας αυτή την οδό και όπως σας είπα θεωρώ την έκθεση εξαιρετική και χαίρομαι που ε, οι ιδέες που περιλαμβάνονται εδώ είναι πάρα πολύ καλές. Ευρωπαϊκή Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σε αντίθεση με άλλους, εγώ διάβασα αυτή την έκθεση και βλέπω πως αρνείται πολλές πραγματικότητες. Πρώτα απ' όλα τα θετικά. Πράγματι πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και η απάτη και να δούμε τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αλλά έτσι σχεδόν παρενθετικά υπάρχει υποψία και διαβάζω από μέσα πως υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση στην περικοπή των μισθών κτλ. Αρνείται τελείως την κριτική που ασκείται στο δούνου του. Και διαβάζω από μέσα οι προγνωστικές, τα προγνωστικά με συγχωρείτε, δεν εκτίμησαν αρκετά την αύξηση της ανεργίας. Επίσης, αρνείται το ότι η όλη κατάσταση δημιουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόβλημα εσόδων και όχι εξόδων και το ότι ε, επιδεινώθηκε πάρα πολύ η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών. Με το λαθασμένο φάρμακο σε όλο και υψηλότερη δόση δεν θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Οπότε πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα φόρος των πλουσίων, δεύτερον η ελεγγύη των κρατών μελών και όχι η ταπείνωση των λαών και κατόπιν ο έλεγχος των λεγόμενων ε, χρηματαγορών, αγορών, επίσης επενδύσεις σε νέες καλές θέσεις εργασίας για τους νέους και άρα ανάπτυξη, πέμπτον να ε, περιοριστεί η φτώχεια των ε, συνταξιούχων αντί να αυξάνεται η ηλικία συνταξιοδότησης και έκτον πρέπει να αναγνωρίσουμε πως αυτά τα οποία γίνονται από το κράτος είναι ανάγκες της κοινωνίας για ε, υπηρεσίες κοινή ωφέλη. Όλα αυτά δεν αναγνωρίζονται. Σας το λέω δηλαδή με τέτοιε εκθέσεις κινδυνεύει η αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωση και οι στόχοι μα για κοινωνική δικαιοσύνη και ίσες ε, ευκαιρίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στόλογιαν παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε οι προτάσεις της έκθεσης του κυρίου Παλώνε σε σύγκριση με την κατάσταση στις χώρες μέλη ενδυναμώνουν την εντύπωσή μας ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Πολλά σκληρά μέτρα έχουν αναλυφθεί από τα κράτη-μέλη για να μειωθούν τα ελλείμματα. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερα μέσα στη διάθεσή της και εργαλεία για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν καλύτερα τα δημοσιονομικά τους με βιώσιμο τρόπο. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τη σημασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που είναι πολύ σημαντικό εργαλείο και πολύ χρήσιμο και αποτελεσματικό. Η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για την σχετική ανάκαμψη που παρατηρήθηκε. Αλλά η πραγματικότητα έδειξε επίσης ότι η ευθύνη του κάθε κράτος μέλους για τα δημοσιονομικά του δεν είναι κάτι που μπορεί να αποφευχθεί. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι πρέπει να θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για το γεγονός ότι ενώ δεκάδες εκατομμυρίων πολιτών της Ένωσης χρειάστηκε να φέρουν το βάρος ε, αυστηρών μέτρων λιτότητας απ' την άλλη διεθνείς εταιρείες πολυεθνικές και ορισμένοι πολίτες διαπράττουν φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή καταφεύγοντας σε φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει και γι' αυτό κάτι να γίνει. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να χαιρετήσω το έργο του εισηγητή και των σκιωδών ε, που ε, παρουσίασαν τόσο επικοδομητικές ιδέες. Οι σημαντικές προσπάθειες ε, που έχουν υλοποιηθεί καρποφόρησαν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τώρα σε θέση με βρία πλουσία να θετήσει την έκθεση αυτή. Αυτός ο συμβασμός αποτελεί εξισουμίωτη πρόοδο στη συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική. Η έκθεση προτείνει ισορροπημένες λύσεις ε, που ε, μακρύνεται από το δόγμα της λιτότητας που χρησιμοποιήθηκε στην Ευρώπη από την έναρξη της κρίσης παρουσιάζονται λύσεις ε, που ε, και κάποιος ρεαλισμός που έλειπε στην Ευρώπη μέχρι τώρα. Ε, τρεις δασκευαστές παρουσιάζονται στην εκθέση αυτή. Η πρώτη ιδέα είναι ότι η ανάκαμψη περνάει και από τις δημόσιες παραγωγικές επενδύσεις και πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος σταθεροποιητής πριν το χάρη μέσα των εθνικών συστηματών συνταξιδότησης. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν μπορεί να υπάρχει δημοσιονομική εξυγίανση διαφορετικά. Δεύτερο, ζητά από την Επιτροπή να δημοσιεύσει τις υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν ε, για να βρει τους πολλαπλασιαστές των ελλημάτων ε, των ε, κρατών μελών. Αν ήταν ακριβείς οι πολλαπλασιαστές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τότε θα μπορούσε να βυθιστεί η Ευρώπη στην ύφεση και γι' αυτό η έκθεση υποστηρίζει ότι μια, φορολογική με μεταρρύθμιση μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πτυχή για την πολιτική εξυγίανση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσφατα παραδέχθηκε τα λάθη του ε, στον υπολογισμό του αντικτύπου της λιτότητας, ε, θα ήταν λυπηρό η Κομισιόν να μείνει μόνη σε δογματικές ε, θέσεις που καθημερινά αμφισβητούνται από την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Ευρώπης. Θέλουμε λοιπόν αυτή η έκθεση να εμπνεύσει τις εργασίες της Κομισιόν καθώς και τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Βεβαίω εύκολα παρακολουθούμε την γραμμή του, αλλά καμιά φορά πρέπει να κοιτάμε και προς τα πίσω για να αντιληφθούμε πώς ε, προέκυψαν τα προβλήματα. Γύρω στο 1973 είχαμε μια κατάσταση όπου όλα τα κράτη ήταν χρεωμένα γιατί βεβαίως ανέμεναν να επανέλθουν οι ε, καλοί καιροί. Και βεβαίως ε, τότε ξεκίνησε ένας πόλεμος υποτίμησης των νομισμάτων για να επιτύχουμε ένα εμπορικό πλεονέκτημα, αλλά βεβαίως τότε τελειώσαμε με την ναι, το ίδιο σημαίνει τώρα με τις φορολογικές μας πολιτικές και μας βλάπτει όλους και βεβαίως αυτό είναι αντίθετο με αυτά τα οποία έλεγε ο Σουμάν γιατί πρέπει να δούμε τα γεγονότα και το τι χρειάζεται η Ευρώπη και οι πολίτες της. Ε, κοιτάμε την Ελλάδα και τα στοιχεία της ανεργίας, η οικονομία καταποντίζεται, τα νούμερα που βλέπουμε είναι τρομακτικά, 56% ανεργία των νέων, και οφείλουμε στους ε, αδελφούς μας Ευρωπαίους να κάνουμε περισσότερα. Σουίμπερν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτό το οποίο λέει η έκθεση του κυρίου Παλώνα και τον ευχαριστώ για τη σκληρή του δουλειά. Πράγματι είναι μια καλή ανάλυση για το πώ μπορούμε να διαχειριστούμε τα δημόσια οικονομικά και ελπίζω να ε, την λάβει υπόψη η κυβέρνηση της Ουαλίας στο τωρινό κλίμα επανεξέταση των δημοσίων οικονομικών, οι κυβερνήσει σε όλα τα επέδα πρέπει να ε, δουν το πού ξοδεύουν τα δημόσια χρήματα. Και βεβαίως αναφέρονται οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, αλλά θα πρέπει και η κυβέρνηση της Ουαλίας να σκεφτεί την δαπάνη δεκάδων εκατομμυρίων ε, ε, ευρώ ή λιρών μάλλον για την εξαγορά του αεροδρομίου του Κάρντιφ όταν δεν μπορούν να το κάνουν εταιρείε ανά τον κόσμο δηλαδή να διαχειριστούν με τρόπο κερδοφόρο ένα τέτοιο αεροδρόμιο πώ θεωρούν ότι μπορούν να το κάνουν αυτό οι υπάλληλοι τη κυβέρνηση τη Ουαλία. ένα αεροδρόμιο μάλιστα το οποίο δεν ε, είναι και ιδιαίτερα δημοφιλές. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ξοδεύουμε τα χρήματα των φορολογουμένων, θα πρέπει να τα επενδύουμε με τρόπο σωστό για να έχουμε δουλειέ και ανάπτυξη.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 Η οικονομική, τραπεζική και χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνει τα τελευταία χρόνια έχει σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά όλων των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σήμερα μια παράλυση στις οικονομικές εξελίξεις και ακόμη και η πολιτική σταθερότητα έχει αποδυναμωθεί σε πολλά κράτη με αρνητικέ προβλέψεις σε ό,τι αφορά την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την αυξανόμενη ανέχεια και ανεργία. Είναι σημαντικό πολιτικέ δημοσιονομική εξυγίανση να λάβουν υπόψη την πραγματικότητα στα διάφορα κράτη-μέλη. Τα μέτρα λιτότητα θα πρέπει να εξισορροπηθούν με μέτρα που να ενισχύουν την κοινωνική προστασία και την κοινωνική ανάπτυξη. Ε, θα πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η έκδοση κοινών μέσων χρέου θα πρέπει να καταστεί πραγματικότητα. Επίση, ε, πρέπει οι νέοι να μπουν στο κέντρο των ευρωπαϊκών λύσεων και να του βοηθήσουμε να συμμετέχουν συμμετέχουν ενεργά στην αγορά εργασία και προκειμένου να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών λύσεων και αυτό το επισημαίνει η έκθεση. Κάθε χρόνο, όχι λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο ευρώ χάνονται λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαπάτης. Επομένως, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να απαντήσουν ε, ηχηρά ε, προκειμένου να βελτιώσουν την ε, εθνική δημοσιονομική κατάσταση αντιμετωπίζοντας αυτά τα φαινόμενα και θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα τους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν εγώ δέχομαι το γενικό ύφο της έκθεσης του κυρίου Παλώνε. Τα περισσότερα κράτη-μέλη χρειάζονται ειδική στρατηγική. Και επομένως πρέπει να βασιστούν σε περικοπές των δαπανών και όχι σε αυξήσεις των φόρων. Επίσης η εξυγίανση σημαίνει δομικές διαμεταρρυθμίσεις όπως πιο ευέλικτες αγορές εργασίας. Ακόμη και η Γαλλία αρχίζει να το κάνει. Όπως δείχνει ο ρόλος που παίζει η οργάνωση των Γάλλων εργοδοτών, το ΜΕΝΤΕΦ. Δυστυχώς όμως υπάρχει πάντα, παραμένει, πολύ μεγάλη, γίνονται πολύ μεγάλες παραχωρήσεις προς την αριστερά και ακόμη πιο σημαντικά το θέμα της εγγύησης για την απασχόληση των νέων μπορεί τελικά να δημιουργήσει περισσότερη ακαμψία στην αγορά. Δεν μπορεί κανείς να υποσχεθεί δουλειές που δεν υπάρχουν και είναι χαρακτηριστική ε, παραμόρφωση των καλών προθέσεων που πολλές φορές εκφράζονται. Τώρα η δια... Δώσω το λόγο στην συνάδελφο Γκάλ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να, συγχαρώ τον κύριο Παλών γιατί εργάστηκε πάρα πολύ καλά στο θέμα της κρίσης και των απαντήσεων στην κρίση. Εγώ συμφωνώ με την διατύπωση πως διαφέρει η κατάσταση από κράτος σε κράτος. Γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε στρατηγικές για την ανάπτυξη που θα οδηγούν σε συγκεκριμένες ανακράτος ε, συστάσεις για να βγούμε από την ε, κρίση. Η εξοικονόμηση βεβαίως είναι κάτι το πολύ βασικό αλλά δεν επαρκεί ε, η λιτότητα από μόνη της. Πρέπει επίσης να αναφερθεί η μείωση των φόρων στην εργασία. Εδώ πέρα υπάρχουν πολλά καλά παραδείγματα και στην χώρα μου, την Ουγγαρία, η Ουγγρική κυβέρνηση ε, έχει αναφέρει πως θα πρέπει να δούμε πολύ ευρύτερα την αλληλεγγύη, να υπάρξει συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους, όχι μόνο περιορισμοί του λαού, αλλά πρέπει και οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες να συμπεριληφθούν εδώ πέρα. Σας συγχαίρω και πάλι εγώ θα υποστηρίξω την έκθεση. <clears throat> Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον εισηγητή όσον αφορά λοιπόν την σταθεροποίηση των ε, προϋπολογισμών. Αυτό είναι βασικό για την ε, διαχείριση των ε, κρίσεων. Αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε πως δεν έχουμε μια ενιαία συνταγή για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μα ακόμα και για την ίδια αρρώστια διαφέρει το φάρμακο ανάλογα με το αν κάποιος είναι παιδί, μεγάλος ή ηλικιωμένος. Οπότε τα αυστηρά αυτά μέτρα που επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν απέδωσαν αυτά τα οποία ελπίζαμε. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε περισσότερα τα κρατημέλη εκείνα τα οποία δεν εφάρμοσαν οπωσδήποτε τη συνταγή του Δουνουτού, όπως παραδείγματος χάρη την Ουγγαρία. ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν υπάρχουν αμφιβολίες ε, στο ότι οι περισσότεροι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, διαφανούν με την πολιτική λιτότητα. Σε αυτό το αποδεικνύει και αυτή η έκθεση ότι δηλαδή η λιτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, μια πολιτική δημοσιονομικής ανάπτυξης. Βλέπουμε ότι επιφέρονται πολύ αρνητικές συνέπειες όπως στη χώρα μου, στην Πορτογουλία, το Κοινοβούλιο ε, εδώ ε, υπερασπίζει τη μείωση της φορολόγησης ε, για τις επιχειρήσεις και τη σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα και αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη μείωση των μισθών, με μεγαλύτερη ενέχεια την απελευθέρωση ε, και την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων ε, επενδύσεων, ε, το, η μείωση των δημοσίων υπηρεσιών και με την επακολούθη άρνηση βασικών δικαιωμάτων στο πληθυσμό. Είναι ηρωνικό οι λύσει που προτείνονται να είναι πάντοτε εμβάθυνση των ίδιων πολιτικών που δημιουργούν το κοινωνικό χάος και εξυπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο Ευχαριστώ Πρόεδρε. το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δημοσιονομικά της Ένωσης για το 2011 και 12 επιβεβαιώνει ότι αυξάνονται τα οικονομικά προβλήματα της Ευρωζώνης. Για να επανέλθουμε στην σταθερότητα είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα, ιδιαίτερα μέτρα λιτότητος και περικοπής των δαπανών, καθώς και η κατάργηση επενδύσεων που δεν αποφέρουν. Με στόχο φυσικά, όπως είπα και πριν, να επανέλθουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα. Απ' την άλλη πρέπει να ληφθούν και μέτρα για τη βελτίωση των φορολογικών εσόδων ώστε να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και την απασχόληση, να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, να αρθούν φραγμοί στη δραστηριότητά τους, αλλά επίσης όλα αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα γιατί οι πολίτες πληρώνουν πολύ ακριβά την έλλειψη αποφασιστικότητάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Ον Λιρέν. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Σας ευχαριστώ εκ νέου για την ουσιαστική συζήτηση που συνάδει με τη σοβαρότητα του θέματος που συζητούμε, γιατί το υψηλό επίπεδο δημοσίου χρέους θα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα, αν όχι το πιο, αν όχι το κυριότερο ζήτημα στην φυστάμενη δεκαετία. Όπως είπα στα εισαγωγικά μου σχόλια, και ως σχολείο της έκθεσης, τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνονται σταδιακά. Και το ίδιο ισχύει και για την εμπιστοσύνη των αγορών στις δράσεις των κυβερνήσεων. Υπάρχει σταδιακή βελτίωση ως προς τις οικονομικές πολιτικές. Φυσικά, η κατάσταση ποικίλει ανάλογα με τη χώρα και γι' αυτό η Κομισιόν ακολουθεί μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για την εξυγίανση, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες ε, προκλήσεις που υπάρχουν σε κάθε κράτος μέλος όταν ε, καθορίζονται οι απαιτούμενες ε, προσπάθειες προσαρμογής. Σε κάποιες από τις παρατηρήσεις σας αναφερθήκατε στο θέμα των πολλαπλασιαστών. Ο κ. Χονγκ τον έφερε νομίζω και κάποιοι άλλοι συναδελφοί σας. Και επίση αναφερθήκατε και στην πρόσφατη μελέτη, στις πρόσφατες μελέτες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η πρώτη ήταν τον Οκτώβριο και μία αναθεωρημένη τον Δεκέμβριο από τον Ολιβιέ Μπρανσόπτα, τον επικεφαλή οικονομολόγο και τον Τανιλή. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το θέμα σύντομα. Καταρχήν, συμφωνούμε με το Διεθνές Ταμείο ότι οι πολυπλασιαστές ε, ε, είναι πιθανό να είναι πιο ψηλοί όταν ε, υπάρχουν δυσκολίες από τα νοικοκυριά. Επίσης συμφωνούμε και κάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι οι πολλαπλασιαστές ποικίλουν ανάλογα με τη χώρα, ανάλογα με το χρονικό διάστημα και ανάλογα με το οικονομικό πλαίσιο. Και από αυτή τη σκοπιά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε τρία ζητήματα όπου η ανάλυση και τα συμπεράσματα του Εθνικού Χρησματικού Ταμείου και της Κομισιόν μπορεί να χάθηκαν ε, σε όλη τη σύγχυση που, προκάλ, που προκλήθηκε σε όλη αυτή τη συζήτηση. Καταρχήν, οι πολλαπλασιαστές ε, αφορούν το αποτέλεσμα της ανάπτυξης της δημοσιονομικής εξυγένσης όπως ε, και της όθησης που δίνεται και η Κομισιόν και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά σε διαφορετικό βαθμό και σε διαφορετικά δείγματα χωρών θεωρούν ότι το πιο σημαντικό ε, πιο σημαντική περίπτωση ε, όπου είχαμε ε, πολλαπλασιαστές για το 2010 πολλές χώρες ε, χρησιμοποιούσαν ε, φορολογικά ε, μέτρα κινήτρων είχαν υποεκτιμηθεί όσο ουσιαστικά η επακόλουθη εξυγίανση πρέπει να πάρει τη μορφή κάποιων μόνιμων μέτρων που θα αντικατοπτρίζονται στην ανάπτυξη. Οι πολλαπλασιαστές αφορούν ε, το αυξητικό αποτέλεσμα της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη θεωρώντας ε, ότι πολλές εξηγιάνσεις μπορεί να οδήγησαν σε ε, ελλείψεις ανάπτυξης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν αναστρέψουμε την εξυγίανση θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης. Και κυρίω ό,τι αφορά χώρε που μπορεί να κινδυνεύουν να χάσουν πρόσβαση στι αγορέ, μια έλλειψη αξιόπιστη εξυγίανση θα οδηγούσε σε τέτοια αύξηση ε, των ασφαλίστρων κινδυνού που ε, τελικά ε, θα έχει καταργήσει οποιοδήποτε όφελος. Ε, ε, οι οικονομολόγοι ερμήνευσαν τα πορίσματά τους ως μια έκκληση να ανατραπούν να οι, οι δημοσιονομικές πολιτικές, να αντιστραφούν οι δημοσιονομικές πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί η Ιταλία το 2011, από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2011. Αν η Ιταλία σε μια κατάσταση όπου ήδη η δημοσιονομική της πολιτική ε, ε ήταν υπορρευματικό, είχε χαλαρώσει περισσότερο τους δημοσιονομικούς στόχους, ε, τότε θα είχαμε σημαντική αύξηση των επιτοκίων που ήταν ήδη υψηλά. Και ουσιαστικά θα οδηγούμασταν ε, σε αδιέξοδο σε σχέση με την κρίση χρέους στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν Πρέπει να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο και το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα γενικό κανόνα για όλες τις περιπτώσεις για τη δημοσιονομική πολιτική. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι το εξής. Υπάρχουν κάποιες αποδείξεις που βασίζονται σε σοβαρή ακαδημαϊκή έρευνα ότι τα επίπεδα του δημοσίου χρέους εμποδίζουν την ανάπτυξη είναι πολύ ψηλά. Τα επίπεδα χρέου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, κυρίως σε ορισμένα κράτη-μέλη, είναι σίγουρα πολύ ψηλά. Έτσι, λοιπόν, είναι το να αφήσουμε το χρέος σε αυτό το υψηλό επίπεδο σημαίνει ότι επίση ε, θα αναχέτιζε την ανάπτυξη. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το δημόσιο χρέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από το 60% περίπου του ΑΕΠ πριν την κρίση πριν 5 χρόνια 60% στο 90% περίπου φέτος και του χρόνου. Και όπως είπα, αναγνωρίζεται βρέως ότι όταν ανεβαίνουν τα επίπεδα δημοσίου χρέους πάνω από το 90% ή το 100% να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική δυναμική και αυτό μεταφράζεται σε μηδενική ανάπτυξη και πολλά έτη. Γι' αυτό αυτό μία προσεκτικά σχεδιασμένη δημοσιονομική εξυγίανση εξακολουθεί να παραμένει απαραίτητη στην Ευρώπη. Και θέλω να κλείσω λέγοντας, επειδή έχει συζητηθεί ιδιαίτερα για το αν θα έπρεπε να έχουμε ονομαστικούς στόχους ή να επικεντρωθούμε σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, είπα στην αρχή των σχολείων ότι έχουμε υιοθετήσει διαφορετική προσέγγιση χώρα για τη δημοσιονομική εξυγίανση και, κάθε, και η προσπάθεια της κάθε χώρας αναφέρεται με συγκεκριμένους διαρθρωτικούς όρους. Αυτό σημαίνει ε, ότι επικεντρωνόμαστε μακροπρόθεσμα στο να μεσοπρόθεσμα στο να μειώσουμε το χρέος και στη ε, διαρθρωτική βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεσοπρόθεσμα ενέχει της ε, απομάκρυσης του αντικτύπου του επιχειρηματικού κύκλου και σημαίνει ότι αν υπάρχει επιδείνωση της ανάπτυξης με έναν απρόσμενο τρόπο, μια χώρα μπορεί να λάβει περαιτέρω χρόνο για να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα, δεδομένου ότι έχει κάνει την απαιτούμενη διορθωτική προσπάθεια. Τέτοιε αποφάσει λήφθησαν πέρσι για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, ας μην ξεχνάμε ότι το επίπεδο του δημοσίου χρέους μας είναι πάρα πολύ ψηλό και γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε με επιμονή προς μια σταθερή εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών μας και για να έχουμε μια υφόρο ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσει εργασία στην Ευρώπη. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Και τώρα ο κύριος Παλαιώνης, ηγητής μας, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο Και επίση ε, να ευχαριστήσω και του και αλλά και του συναδέλφου που πήραν το λόγο σήμερα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Εγώ έχω μια προσέγγιση συγκεκριμένη. Κανείς δεν γνωρίζει την πλήρη αλήθεια, επομένως είναι δύσκολο το έργο μου. Άκουσα μια σειρά συναδέλφων ε, που μίλησαν και έκαναν κάποια ενδιαφέροντα σχόλια και έχουμε και μια σειρά τροπολογιών που προτάθηκαν ε, και μέσω συμβεσμών έγιναν δεκτέ. όμως έχει δίκιο ο ε, δεν μπορούμε να φυσικαζόμαστε γιατί δεν έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Το αντίθετο, εξακολουθεί να είναι ανοιχτή συζήτηση και υπήρξαν ε, και κάποιες κριτικές γιατί χρησιμοποιήθηκε όρος ιατρική για την αρρώστια. Όμως ας είμαστε προσεκτικοί γιατί όταν κάποια προβλήματα αντιμετωπίζονται χωρίς τη δέουσα επιμέλεια είναι κακή και ιατρική. Ακούσαμε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση εξακολουθεί να είναι ένα ανοιχτό ζήτημα. Ο τρόπος που πρέπει να υλοποιηθεί είναι ένα ανοιχτό ζήτημα προς συζήτηση. Κανένας ε, δεν γνωρίζει ποια είναι η πανάκια έχουμε διάφορες σχολές ε, σκέψης που αναδύονται και από τον ακαδημαϊκό κόσμο και ε, πρέπει να βρούμε ποιο είναι το σωστό μείγμα μεταξύ φορολόγησης και περικοπής των δημοσίων δαπανών. Δεν υπάρχει μία συνταγή που να ταιριάζει σε όλους. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών που μας επιβάλλουν να αντιμετωπίσουμε τι καταστάσει ανάλογα με την ιδιαιτερότητα τη κάθε χώρας. Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα είναι χώρε του Νότου, αλλά η κατάστασή τους είναι εντελώ διαφορετική. Εγώ τι ζητώ κύριε Επίτροπε να ε, έχουμε ένα ανοιχτό διάλογο για να προχωρήσουμε και το πραγματικό πρόβλημα που πρέπει να συζητήσουμε είναι ένα διώνυμο, δηλαδή να έχουμε την εξυγίανση και την ανάπτυξη και πρέπει να μιλάμε και για ανάπτυξη και για δημοσιονομική εξυγίανση. Δεν, αν δεν θέσουμε και την ανάπτυξη μέσα στη συζήτηση, τότε διακινδυνεύουμε να μπούμε ε, σε ένα φαύλο κύκλο μεταξύ του προβλήματος των δημοσίων δαπανών και του προβλήματος της ύφεσης για αυτό το θέμα, εγώ νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε ε, και να βάλουμε σε πρώτη θέση το συμφέρον των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Παλώνα. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε. Η ψηφοφορία για την έκθεση του κυρίου Παλώνα θα διεξαχθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων. Και θέλω πρώτα να δώσω το λόγο στον συντάκτη της προφορικής ερώτησης, τον συνάδελφο Σάντσες Πρεσέντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.